Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Την προσοχή σας παρακαλώ. Ξέρετε, λαμβάνει χωρί ολομέλεια. Και έχουμε και ένα σημείο τώρα της ΛΥΜΠΕ που συζητείται αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια και βρισκόμαστε εμείς εδώ για μια ψηφοφορία. Επομένως, σας είμαστε γρήγοροι. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι κάθονται, τουλάχιστον ε, όσο κάθεστε, επιτρέψτε μου να κάνω τις ε, ανακοινώσεις. Έγκριση της ημερησίας διάταξη. Αναβάλουμε μία ψηφοφορία για την γνωμοδότηση Λίβεν για την Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι το ένα. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Εγκρίνεται. Δεύτερον, γλωσσικό προφίλ. Διαθέτουμε όλες τις γλώσσες εκτός από μαλτεζικά, ε, αρχαιρλανδικά, κροατικά και λετονικά. Καθίστε ησύχως παρακαλώ. Πρέπει να εγκρίνουμε τις συστάσεις των συντονιστών. Διορισμός των εισηγητών για γνωμοδοτήσεις. Ναντίν Μωράνο, εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Θέλετε το μικρόφωνο. Thank Actually, she did the... Έκανε το σωστό. Παρακαλώ. Λίγη ησυχία, παρακαλώ. Θα είμαστε ταχείς, γιατί συζητείται ένα σημείο λίμπε στην ολομέλεια αυτή τη στιγμή. Να είμαστε γρήγοροι, παρακαλώ. Στη συνέχεια, ο Ντρακοβάρη και είναι εισηγητή για την τεχνητή νοημοσύνη ε, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στα οπτικοκουστικά. Συμφωνείτε? εγκρίνονται οι διορισμοί αυτοί. Κατόπιν, κατά εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, έχουμε το πρόγραμμα για τις λύσεις διαλειτουργικότητας και τα κοινά πλαίσια σε σχέση με την κατανομή των δαπανών για το 2020. Κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της ε, ΛΥΜΠΕ μέσω του newsletter στις 10 Ιανουαρίου. Και η εσωτερική προθεσμία για αντιρρήσεις είναι στις 20 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Εντάξει. Αν συμφωνείτε, τότε μπορούμε να περάσουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία και πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πριν, την ηλεκτρονική ψηφοφορία έχουμε ένα ουσιαστικό σημείο που είναι η πρόταση κανονισμού που καταργεί την απόφαση του Συμβουλίου είναι το σύστημα VIS. Δίνουμε ε, εντολή στη διαπραγματευτική ομάδα να ξεκινήσει διαπραγματεύσει σε τριμερεί διαλόγου. Δύο τριμερεί διαλόγοι έλαβαν χώρα. Ο πρώτο 28 Νοεμβρίου. Έχουμε τον εισηγητή εδώ, τον συνάδελφο κ. Ρανζέλ. Σας ευχαριστούμε που θα μας εξηγήσατε τι γίνεται πριν να περάσουμε στις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τον περασμένο Οκτώβριο αρχίσαμε τις εργασίες στο φάκελο αυτό. Θα έλεγα ότι ακολουθούμε ένα σταθερό ρυθμό παρά διάφορα εμπόδια. Και παρόλα αυτά Θέλω να υπογραμμίσω το επικοδομητικό πνεύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη Φιλανδική Προεδρία. Ήταν αξιοσημείωτη και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να πούμε το ίδιο και για την Κροατική Προεδρία. Σε λιγότερο από έξι μήνες. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατό να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο και ότι θα έχουμε τελικά ένα ενισχυμένο σύστημα ΒΙΣ, πληροφόρηση των Επί της ουσίας, νομίζω ότι σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο, όμως ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε συμβιβασμό για κάποια από τα θεμελιώδη ζητήματα για το Κοινοβούλιο. Καταρχήν, τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων, ιδίως ε, για τα παιδιά με μεγάλες ασφαλιστικές δικλείδες μπορούν να εισαχθούν σε σύστημα πληροφορικής. Δεύτερον, την ενίσχυση αρχιτεκτονικής συστήματος ΒΙΣ. Τρίτον, την ενίσχυση των ε, μηχανισμών υποβολής αναφορών και την προθεσμία το μέγιστο δύο έτη για να έχουμε ε, ένα νέο ΒΙΣ που να λειτουργεί. Και τέλος, να έχουμε κατάλληλους ελέγχους σε άλλα συστήματα που θα σέβονται την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα και χωρίς ε, να μπλοκάρουν την λειτουργία των υπόλοιπων συστημάτων. Έτσι λοιπόν και κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ε, έχουμε κρεμεί θέματα από την προηγούμενη θητεία. Όλα ε, τα μέλη είναι νέα για το φάκελο αυτό. Έτσι λοιπόν οι συνάδελφοι σε αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικοί και μαζί έχουμε μπορέσει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και κλείνω τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο τους. Έτσι έχει η κατάσταση σήμερα. Thank you for your short σας ευχαριστώ κύριε Ρενζέλ, για τη σύντομη παρουσίαση. Οι σκιώδεις, ε, αν θέλουν, μπορούν να πάρουν το λόγο. Έχουμε τον κύριο Τσουλάρου για τους ασοσιαστές και τον κράτες, τον κύριο Τουντοράκε από το Ρινιού, σχόλια. Όχι. Άλλη και. για τους πράσινους. Όχι. την κυρία Νικοσόνοβα από το ECR και την κυρία Ντάλη από την ΚΟΕ. Αφού κανείς δεν λέει κάποιο άλλο, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ήταν πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Δώσαμε μια καλή μάχη και θέλω να τον ευχαριστήσω και για το έργο του. Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να προχωρήσουμε αμέσως στις ψηφοφορίες. Ευχαριστούμε κύριε Ρανζέλ. Ολοκληρώνεται το σημείο αυτή. Ας περάσουμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχουμε κάποιες ψηφοφορίες. Σας είμαστε ταχύς.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 just watch. Colleagues. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, παρακαλώ την προσοχή σας για ένα λεπτό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στι 7 ε, και 20 έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία, οπότε καταλαβαίνω οι συνάδελφοι είναι εδώ, αλλά αν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε. Θα ήταν πρόβλημα για να κερδίσουμε κάποια λεπτά και να επιστρέψουμε το συντομότερο στην Ολομέλη. Αν συμφωνείτε, ωραία, πάμε. Okay. So, somebody will... Okay, first. We... Παρακαλώ. σε τεφά την απαλλαγή για την εκτέλεση του προπολογισμού των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων για το οικονομικό έτος 2018. Η κυρία Μέτσολα είναι η συγγήτρια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτήν την ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν δουλεύει. Για μένα τουλάχιστον όχι. Δεν ξέρω για σας. Excuse me. Let me change. Let me change the card to see. Για να αλλάξω κάρτα να δω. Now, now it works. Α, εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Για να δούμε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τι είπατε, ψηφοφορία, συγγνώμη, τροπολογία 4. Την έχετε. Υπάρχουν προβλήματα. Τροπολογία 4. Εντάξει, ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Διορθώνει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 8. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε στο κείμενο όσο έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία. Πέρας. Έγκρινεται. Ευχαριστούμε. Πάμε στο δεύτερο φάκελο. Απαλλαγή της ε, Europol για το 2018. Και πάλι, γύτρα κυρία Μέτσολα. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα στο τελικό κείμενο όσο έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ευχαριστούμε κυρία Μέτσολα και πάλι εγκρίνεται. Πάμε στο επόμενο. Έκθεση απαλλαγή της κυρίας Μέτσολα για τη ΣΥΠΟΛ. Και πάλι το 2018. Τροπολογία 1. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολόγια 2. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα στο κείμενο όσο έχει τροποποιηθεί, τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Ωραία, και πάλι εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Πάμε στην επόμενη έκθεση απαλλαγή για την Eurojust και πάλι το 2018. Ξεκινάμε. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 10. Άρχεται. Α, όχι. 9. Καταπέμπτη. Επειδή εγκρίθηκε η συμβαστική 4 της ε, συνολικής νομοδότησης για, τους, ε, για τα θεσμικά όργανα. Επομένω, αυτή η τροπολογία 9 καταπίπτει. Πάμε στην ε, τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τελικό κείμενο, όσο έχει τροποποιηθεί. Πάμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η επόμενη έκθεση είναι επίσης της κυρίας Μετζόλα. Πρόκειται για την απαλλαγή για το 2018 EU Λίσα. Τροπολογία 1. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται με μία διαφορά. Τροπολογία 2. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Αρχή. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Ναι. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται 11. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία αρχή. Τέλος. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Η επόμενη απαλλαγή αφορά το EDPS, ε, Εποπτική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων, τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται 2. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίθηκε και αυτή. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την ψηφοφορία για την ΦΡΑ, Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 2018 απαλλαγή, η κυρία Μετσόλα είναι Είναι η τιμητική της βραδιά σήμερα. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Συμβιβαστική τροπολογία 1, αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, αρχή της ψηφοφορίας. 4. υπόλοιπες καταπίπτουν. Τέλος. Εγκρίνεται η 4. 5. Ψηφίζουμε την 5. Αρχή. Τέλος. Εγκρίθηκε. 6. Τροπολογία 6 ψηφίζουμε. Τέλος. 7. Εγκρίθηκε η 6. Τροπολογία 7. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται 7. 8. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται 9. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 10. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται και αυτή. Συμβιβαστική 2. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 14 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε το τελικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας, τέλος. Εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε την κυρία Μετσόλα. Και τώρα προχωράμε στην απαλλαγή της ε, Frontex. 2018 τροπολογία 1 ψηφίζουμε τέλος εγκρίνεται 3 ψηφίζουμε τέλος απορρίπτεται 4 Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην συμβιβαστική 1. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 14. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 15. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 16. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. εγκρίνεται. Τροπολογία 20, αρχή. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5, αρχή. Τέλος ψηφοφορίας. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας από το ΕΛΚΑ υπεράριθμος. Κυρία Ζητόφσκη. Εγκρίνεται η 16. Και τώρα περνάμε στην 25 τροπολογία. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Το κείμενο τροποποιημένο. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίνεται. Απαλλαγή. την άζω. Για το 2018. Πάρει η συγκήτρια είναι η κυρία Μετσόλα. Συμβιβαστική 1. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίθηκε. 5. Ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην συμβιβαστική 2. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 10. Αρχή. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. 11. Αρχή της ψηφοφορίας. Τροπολογία 11. Εάν είχε υιοθετηθεί η 10, θα είχε καταπέσει. Αλλά απορρίψαμε τη 10. Οπότε ψηφίζουμε την 11. Τροπολογία 11. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 3. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίθηκε. 15 αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εγκρίθηκε. 16. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. 4. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική, ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Ευχαριστώ την κυρία Μετσόλα. Πάμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε το παρατηρητήριο για τα ναρκωτικά και την για το 2018. Και πάλι η κυρία Μετσόλα, συγγητρία, τρεις τροπολογίες. Τροπολογία 1, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 2, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται τροπολογία 3, έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Και έχουμε το τελικό κείμενο που τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λήξη. Εγκρίνεται. Και έχουμε και μια ακόμη απαλλαγή για την εφαρμογή του Γενικού Προπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 για τις εκτελεστικές υπηρεσίες της Επιτροπής. Η κυρία Μετσόλη Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Έναρξη. Τροπολογία 2. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. 4. Έναρξη. Λήξη. 5. Έναρξη. Συγγνώμη, εγκρίνεται η 4. 5. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Γιατί η 7 καταπίπτει. Άρχεται η ψηφοφορία για την 8 λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία για το κείμενο πως τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λήξη. Εγκρίνεται. Και τελειώσαμε. Ευχαριστούμε την κυρία Μετσόλη. Σας ευχαριστώ όλους. Τόσο αστείο, κύριε Φώστα. Ήταν γελίο. Πραγματικά ήταν τόσο αστεία αυτή η ψηφοφορία για τις απαλλαγές. Τόσο γελία.